Right. Good Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε όλοι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημείο 2 στη μερίσια διαταξή είναι η έγκριση αυτής. Σχόλια έχετε? Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διαταξή. Σημείο 3. Ανακοινώσει του Πρόεδρου δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Σημείο αριθμών 4. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Έχουμε τα πρακτικά της συνεδρίας 13 Νοεμβρίου 2017. Αν δεν έχετε σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίας θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Και ερχόμαστε τώρα στα σημεία 5 και 6. Είναι κοινή ανταλλαγή απόψεων συζήτηση και για τα δύο σημεία και θα ήθελα να καλωσορίσω τους συμμετέχοντες στην ε, δημόσια ακρόαση. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Μαρίτσια Σχάκε. Καλώς όρισες Μαρίτσια. Σύντομα να σας αναφέρω το θέμα. Πρόσφατα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρηση ενδιάμεση για τα νέα χρηματοδοτικά μέσα εξωτερικά ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Η παρούσα έκθεση φιλοδοξεί στο να ακουστούν οι απόψει μα στην προετοιμασία τη επόμενη νομοθεσία. Ωστόσο, αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει με την συνήθι νομοθετική διαδικασία που είναι στην απόφαση ε, όπως έγινε και για την τρέχουσα περίοδο. Σήμερα τι θα κάνουμε, έχουμε προκαλέσει ε, υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπής και εκπροσώπου ε, τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να μα δώσουν ενημέρωση για τα βασικά σημεία και να κάνουν προτάσει ε, πολιτική και συστάσει για να τι λάβουμε υπόψη. Ένα από τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες που έχουν οριστεί. Ωστόσο, έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στο γενικό πλαίσιο σχετικά με την παροχή βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν λοιπόν οι ε, εκπρόσωποι γιατί δεν έχουν καταθέσει κάτι εξοδότηση πράξης επιπλέον η ΑΦΕΤ θα συζητήσει και με την κυρία Μογκερίνη και τον κύριο Χάν αυτή τη στιγμή ε, γίνουν οι προτάσεις για το 18 με 20, μάλλον 21 και 22 Φεβρουαρίου, αυτό ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Επιτροπή Εξωτερικών επίσης έχει ε, ιδρύσει και μια ομάδα εργασίας με προεδρία της κυρίας Χάκε ε, για τον έλεγχο της λειτουργίας και της εφαρμογής αυτής ε, της διαδικασίας το 2014. Συμμετέχει και στην προετοιμασία των στρατηγικών διαλόγων. Θα ήθελα να σας συστήσω τώρα τους προσκεκλημένους μας. Γνωστός και μη εξαιρεταίος και τακτός επισκέπτης μας είναι ο κύριος Κρίστια Λέφνερ, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τη ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Τον συνοδεύει ο κ. Φιλιμπέρτο Τσεριάνη Σεμπρεγκόντι, επικεφαλής ε, της ε, υπηρεσίας Συντονισμού Αναπτυξιακή συνεργασίας Είναι η κυρία Μίριαμ Φεράν, ε, Διευθυντή για τη Στρατηγική και την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Χίλτε Χάρτεμαν, Διευθύντρια των Χρηματοδοτικών Μέσων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Ζαν Λουί Βίλ είναι αυτή τη στιγμή διευθύνων το People and Peace στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Ο κύριο Άντρου Σέριφ επικεφαλής του προγράμματος εξωτερικής δράσης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο του Μαστρίχτ και η κυρία Ισαμπέλη Ιωαννίδη, αναλύτρια πολιτική στην υπηρεσία, την ερευνητική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα μας παρουσιάσει την αντίστοιχη μελέτη που έχει γίνει για το θέμα. Ο κύριος Γκίρτσαρτ Γιάνγκς από το Carnegie Europe θα μας παρουσιάσει κάποιες μελέτες από την Τουρκία, Ουκρανία και Αίγυπτο και τέλος είναι η κυρία Σόνια Ρένες Τζιβανίδη, εκτελεστική διευθύντρια του ΕΠΛΟ, European Peace Building Liaison Office, Βρυξέλλες. Πώς θα το διοργανώσουμε. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Σχάκε που θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της, το σχέδιο έκθεσης για ένα πεντάλεπτο περίπου και θα ήθελα να δώσω στο καθένα από τους τέσσερις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, Πέντε λεπτά για τα σχόλιά τους και σε επτά λεπτά. Και μετά ε, θα γίνει μια συζήτηση και θα ακούσουμε και τους κοιόδης ηγητές για μισή ώρα. Ε, θα κλείσει ε, στη συνέχεια η κυρία Σχάκε που θα προεδρεύσει μάλιστα και θα κάνει τα καταληκτικά και συμπερισματικά σχόλια. Αυτά από πλευρά μου το λόγο έχει η συγκεκριά. Σε ευχαριστώ πολύ Ντέβιτ, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το σχέδιο της έκθεσης και την ενδιάμεση αναθεώρηση σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά οικονομικά εργαλεία. Μιλάω όχι μόνο ως εισηγήτρια, αλλά και ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας, στην οποία είστε όλοι καλοδεχούμενοι για να πάρετε μέρος στον έλεγχο των δημοσίων πόρων που δαπανούμε σε εξωτερικές δράσεις. Οι παρατηρήσεις μου βασίζονται στις εμπειρίες που αναπτύξαμε στην ομάδα εργασίας με το στρατηγικό διάλογο, τις προετοιμασίες για την ενδιάμεση αξιολόγηση, τις εξωτερικές αξιολογήσεις, τις συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους και τα μετά που αφορούν την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ελπίζουμε ε, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με την έκθεση αυτή στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του 2020. Τι μάθαμε από όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό με τα οικονομικά εργαλεία να έχουμε συνοχή και στρατηγική αντιμετώπιση, να επιδεικνύουμε ελαστικότητα όταν αλλάζουν τα πράγματα, αλλά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για λιγότερη κρατία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτήρια αξιολόγηση στις πολιτικές για να μπορούμε αργότερα να καταλάβουμε κατά πόσον έχουμε επιτελέσει τον προορισμό μα. Έχουμε επιτυχεί του στόχου μα και να οργανωθεί με έναν καλύτερο τρόπο έλεγχο από το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι το όλο πλαίσιο με τους στρατηγικούς διαλόγους δεν είναι ικανοποιητικό. Πολύ συχνά υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης ή ε, έρχονται καθυστερημένα οι πληροφορίες ε, δεν δίνουμε την εντύπωση ότι διεξάγεται ένα σοβαρό στρατηγικό διάλογο. Δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν συγκρούσει. Αυτά σε ό,τι αφορά το όλο πλαίσιο. Δεν θέλω να υιοθετήσω μία δογματική στάση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερος έλεγχος, περισσότερο στρατηγικές δράσεις και διαφάνεια προς τους εταίρους μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μας καθορίζουν οι πολιτικές και όχι τα μέσα και θα πρέπει να φροντίζουμε έτσι ώστε <clears throat> θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ε, θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Η νέα προτεραιότητα είναι η διαχείριση και το να ε, δίνουμε πόρους προς τα εκεί, ενδεχομένως είναι εις βάρος άλλων πολιτικών στόχων και αυτά συμβαίνουν χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος. Σκέφτομαι την Τουρκία, σκέφτομαι τα διάφορα καταπιστεύματα Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις λείπει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Μολονότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων, όπως σας είπα δεν νομίζω θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία δογματική στάση, δεν θα πρέπει να προσκοληθούμε σε μέσα απλά και μόνο επειδή υπάρχουν, θα πρέπει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα που αφορά τη διακυβέρνηση. Το ερώτημά μου λοιπόν στους εκπροσώπους της Επιτροπής και των Εξωτερικών Υπηρεσιών είναι τι μορφή θα προσλάβει αυτή η διακυβέρνηση, πώς θα έχουμε την βεβαιότητα ότι σε μια μελλοντική αρχιτεκτονική η οποία θα καταλήξει σε ένα πάντρεμα ε, διαφόρων τομέων, πώς ε, ο συντονισμός, τι μορφή θα προσλάβει ο, συντονισμός και ποιος θα είναι ο μελλοντικός ρόλος του Κοινοβουλίου. Γιατί αν για κάποιο λόγο υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, υπάρχει ο κίνδυνος να μπει στο περιθώριο το κοινοβούλιο και αυτό πιστεύω ότι θα ήταν απαράδεκτο και θα υπάρξουν πολλές αντιστάσεις από εσά. Αυτές είναι οι αρχικές μου παρατηρήσεις από την ομάδα εργασίας και πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Ε, είμαστε υπόλογοι για κάθε ευρώ που δαπανάμε. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε, να τιμήσουμε όχι μόνο τους εταίρους μας, αλλά και τις αρχές που πρεσβεύουμε. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε σε αυτούς που συμμετέχουν στο πάνελ. Ο κύριος Λεφλέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας προς τον ίδιο και τους συναδέλφους μου. Να ευχαριστήσω τη Μαρίζα Χάκε για την δουλειά την οποία έχει ήδη κάνει. και τα στοιχεία τα οποία μας έχει προσφέρει για συζήτηση σήμερα. Δεν θα περάσω τώρα σε πάρα πολλές λεπτομέρειες της ενδιάμεσης αναθεώρησης γιατί στο τέλος του μήνα θα υπάρξει μια συνάντηση σε επίπεδο στρατηγικού διαλόγου με την ΑΦΕΤ και αργότερα με την ΤΕΒΕ για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Θα σχολιάσω λίγο αυτά που είπε η Μαρίζα. Να δούμε τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από τις εμπειρίες που είχαμε μέχρι τώρα και να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε καλύτερα την επόμενη γενιά των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων. Θα συμφωνήσω με τις βασικές ιδέες που συμμορφήσε η Χάκε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε στρατηγικά, ευέλικτα, με σωστά κριτήρια αξιολόγησης και με πραγματικό έλεγχο από το κοινοβουλευτικό σκέλος, όπως και καθοδήγηση από τα κράτη-μέλη να δούμε πώς θα το πετύχουμε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να υπογραμμίσω πέντε συμπεράσματα στα οποία νομίζω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε με τα προγράμματά μας μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα. Πρώτον, θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε μια συνολικότερη αντίληψη για το, για το τι θέλουμε να πετύχουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, να τα δημοσιοποιούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πολλούς από τους τομείς της πολιτικής και πολλές από τις προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται από πλευράς μας διασυνδέονται μεταξύ τους ας πούμε είναι προφανής ε, η σχέση ανάμεσα στη μετανάστευση από τη μία και την ασφάλεια από την άλλη. Δεν μπορούμε απομονωμένα να τις αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αίτια τα οποία οδηγούν στην τρομοκρατία, να δούμε ε, τι ακριβώς έχει οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς να μεταναστεύσουν είτε ε, εθελοντικά είτε υποχρεωτικά, αναγκαστικά και να προσπαθήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία να μας δώσουν τα σωστά συμπεράσματα. Ένα δεύτερο μάθημα που πήραμε είναι ότι για να έχουμε την σωστή ανταπόκριση στις ρευστές πολιτικές συνθήκες και αλλαγές απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι να απλοποιήσουμε τις δομές που χρησιμοποιούμε και να απομακρύνουμε κάποια από τα εμπόδια που έχουν φράξει μερικές φορές τις διαδικασίες τα τελευταία χρόνια. Ήδη από το 2014 βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην παρούσα σχεδίαση των προγραμμάτων μας που δεν μας επέτρεψαν να είμαστε επιτυχείς όσο γρήγορα το επιθυμούσαμε ε, τιμώντας τις πολιτικές μας υποχρεώσεις, τις ανηλυμένες πολιτικές μας υποχρεώσεις. Να δούμε πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές και προσφυγικές ροές και στα πλαίσια της δύσκολης διαδικασίας μετακίνησης των πιστώσεων ανάμεσα στους διαφορετικούς τίτλους και θέσεις του προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να εμφυσίσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα μέσο ή στα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι καθοριστική πρόκληση για μας. Στο ίδιο επίπεδο, τα πολλαπλά προγράμματα για κάθε μέσο μας εμποδίζει και εμάς σαν Επιτροπή και σας σαν Κοινοβούλιο να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα των δράσεων αυτών και με την εικόνα αυτή να σχεδιάζετε τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε. Μια απλοποιημένη αρχιτεκτονική, μια πιο απλή δομή θα μας επιτρέψει να δώσουμε πιο συνεκτικές απαντήσεις σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και με περίπλοκο τρόπο όλο και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να ομαδοποιήσουμε τα διάφορα μέσα, διατηρώντας όμως ε, κάποιους θυλάκους ε, ε, θεματολογικούς και γεωγραφικούς έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα διασφαλίσουμε μια διαδικασία απλούστερη αλλά από την άλλη η σωστή πολιτική στόχευση θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε πάντα την προσοχή μας τραμμένη σε συγκεκριμένους επιλεγμένους τομείς σε σχέση με όλες τις αλλαγές που συντελούνται. Ένα τρίτο συμπέρασμα ή μάθημα, όπως είπε και η κυρία Σχάκε, θα πρέπει η πολιτική μας να ακολουθεί ακριβώς πολιτικές αρχές και όχι να επιβάλλεται από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα μας αποτρέπει από το να έχουμε μια πλήρη και συνολική εικόνα και αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε και μέσα από την ενδιάμεση αναθεώρηση η διέρεση ανάμεσα σε διαφορετικά μέσα, η γεωγραφική αναχώρα διέρεση μας κάνει να ξεχάσουμε τη συνολική εικόνα. Βλέπουμε τα δέντρα αλλά δεν βλέπουμε το δάσος. Απαιτείται λοιπόν στα πλαίσια των πολιτικών εξελίξεων, των διαλόγων και των μορφών ελέγχου να μην πέσουμε στην παγίδα να μας επιβάλλουν την πολιτική μας τα διαθέσιμα μέσα. Ε, μέσα τα οποία επιβάλλουν με διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές πορείες, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται μέσα σε ένα ευέλικτο πλαίσιο. Περνώ τώρα στο τέταρτο συμπέρασμα μάθημα. Μεγαλύτερη ευελιξία. Μεγαλύτερη ευελιξία δεν σημαίνει μικρότερος έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίθετα, Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευελιξία θα σας δώσει και εσάς καλύτερες δυνατότητες ελέγχου των στρατηγικών μας προοπτικών. Προσπαθούμε και εμείς να δημοσιονομήσουμε σε εισαγωγικά όλα αυτά τα ε, επιπλέον ταμεία και καταπιστεύματα, σε συνεργασία βέβαια μαζί σας Θέλουμε επίσης ε, να υπάρξουν μηχανισμοί που θα διασφαλίσουν τις ικανότητες του Κοινοβουλίου να ασκήσει σωστά την κοινοβουλευτική του ελεγκτική διαδικασία και να κρατήσουμε την διαφάνεια που απαιτείται σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε και τελευταίο μάθημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις επιτυχίες τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα αλλά και να καλύψουμε τα κενά τα οποία είναι απαραίτητα για την πολιτική επιτυχία. Να χρησιμοποιήσουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αηφόρο ανάπτυξη και τα επόμενα στρατηγικά αναπτυξιακά μέσα έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις καινοτόμες χρηματοδοτικές διαδικασίες ε, για τα προγράμματά μας. Ταυτόχρονα στον τομέα της ασφάλειας Είναι προφανές ότι όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω του, του κοινοτικού προϋπολογισμού γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας εξαιρεί κάποιες ε, παρεμβάσεις αλλά σαν παράδειγμα η επέμβηση στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ειρηνευτικής ε, του ε, Ευρωπαϊκού Ειρηνευτικού Μηχανισμού ή μέσου είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο στρατιωτικό εάν χρειαστεί. Απαιτείται λοιπόν η κατάλληλη προσαρμοσμένη εργαλειοθήκη για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και είναι σαφές ότι οι δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμβατες με τις τρέχουσες δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό και με τις υποχρεώσεις τις οποίες συλλογικά έχουμε αναλάβει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικής δράσης. Συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Λέφνα. Η Ευχαριστώ. Η κυρία Φεράν Εγώ θα περιοριστώ στο να κάνουμε μια καταγραφή-απογραφή ε, των δύο μέσων που έχουμε στην αρμοδιότητά μα το προενταξιακό και το μέσο για τη γειτονία. Θα σας δώσω τα βασικά ευρήματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης, ε, που τα κυριότερα έχουν βρει στην έκθεση της κυρίας Χάκερ. Από τη γειτονία, σύμφωνα με την ε, διάμεση αναθεώρηση εξυπηρετεί το σκοπό του. Στόχο είναι να εφαρμοστεί ανανεωμένη πολιτική γειτονία και με ευελιξία να αντιδρούμε σε μικρέ κρίσει που είχαμε πολλέ. Ουκρανία, την Ισία, η μεταναστευτική και άλλε, για να σα αναφέρω κάποιε ενδεικτικά. Η εφαρμογή τη αρχή διαφοροποίηση επίση ε, είναι πολύ σημαντική γιατί ε, ε, προσαρμοζόμαστε στις κειμενόμενες ε, και ποικίλε ανάγκες των κρατών μελών. Έχουμε επίσης δοκιμάσει και το πώς μπορεί να αντιδρά αυτό το μέσο σε διάφορες μικρές κρίσεις που αντιμετωπίσαμε στην περιοχή και αυτή η ευελιξία Ακόμα και αν χρησιμοποιείται πάρα πολύ χρήσιμα και με τα δύο καταπιστεύματα που έχουν ε, δημιουργηθεί, αγγίζει τα όρια της. Η κρίση και η πρόληψη των κρίσεων είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας, όπως είπε και ο Κρίστιαν, όταν σχεδιάσουμε τα νέα μέσα. γιατί. Αποτελεσματικότητα επίσης έχει βελτιωθεί το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα σε διάφορες γειτονικές χώρες, σταθεροποιώντας ε, χώρες όπως η Ορδανία, την Ισία, Ουκρανία. Επίσης, όπως σημειώνεται στην έκθεσή σας, το πολιτικό πλαίσιο σε πολλές χώρες δεν ε, βοήθησε να γίνουν ε, μεταρρυθμίσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και χρηστή διαχείριση. Στο νέο λοιπόν ENI ε, θέλουμε να προωθήσουμε τη σταθεροποίηση της δημοκρατίας και τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες που έχουν δεσμευτεί να το πράξουν. Δηλαδή είναι πιο ε, μεικτό το τοπίο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποτελεσματικότητα, η διάμεση αναθεώρηση εντόπισε κάποια ε, θέματα, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται επιτυχώς με αποδεκτό κόστος για τις λειτουργικές διοικητικές δαπάνες. Είχαμε έγκαιρη παρέμβαση και ε, επίσης οι νέοι τρόποι ε, μεικτής το λεγόμενο blending, συνδυασμό χρηματοδότηση από διάφορους πόρους, βοήθησαν γιατί κινητοποιήθηκαν επιπλέον πόροι. Η ενδιάμεση αναθεώρηση επίσης έδειξε ότι τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης δίνουν ε, σωστά πληροφορίες. Βεβαίως χρειάζεται να αναθεωρηθούν, αυτό θα πρέπει στο μέλλον να το συζητήσουμε για τη μελλοντική εφαρμογή ε, των ίδιων μέσων των χρηματοδοτικών της επόμενης γενιάς. Επίσης προβλέπεται αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με την υποβολή εκθέσεων. Σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία, το μέσο έχει αποδειχθεί ότι παρέχει προστιθέμενη αξία, δίνει σταθερότητα, ε, ουσιαστική χρηματοδότηση από ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο με διάφορους τρόπους και υπάρχει δυνατότητα συντονισμού και κινητοποίησης πραγματογνωμοσύνης από τα κράτη-μέλη και διαμόρφωση της πολιτικής ε, με διάλογο με τις διάφορες εθνικές αρχές. Επανέρχομαι στην εισαγωγή. Έχει αποδοχθεί ε, χρήσιμο και καλό. Εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το μέσο για τη γειτονία. Και είναι και ιστορική ευκαιρία τώρα να συνεργαστούμε με τους γείτονες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπως αναφέρεται στην ε, συνολική στρατηγική. Έρχομαι τώρα στο προενταξιακό μέσο, το ΙΠΑ. Και αυτό θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί το σκοπό του σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την επερχόμενη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα δώσει μια πλατφόρμα για ακόμα μεγαλύτερη ολοκλήρωση χάραξη πολιτικής και οικονομικής ενίσχυσης. Επίσης έχει υποδεχθεί πολύ ευέλικτο και μάλιστα ε, όταν είναι επιτακτικές ανάγκες και επίγουσες. Ας πούμε, το μεταναστευτικό, η προσφυγική κρίση, η απόκριση που δώσαμε και στο ΙΠΑ, το προεταξιακό μέσο, καταφέραμε να υποστηρίξουμε τα Δυτικά Βαλκάνια και τη διευκόλυνση ε, για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Εστιάζει πάρα πολύ στις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στο πρωταξιακό μέσο, χάρη στην εισαγωγή μιας προσέγγισης που λέγεται τομεακή πλέον. Ακόμα και είναι σε πρώιμα σε στάδια εφαρμογής, ε, θεωρείται σημαντικό. αν και τα κονδύλια περιορίζονται σε λίγους τομείς, στα θεμελιώδη όπως ονομάζονται στη στρατηγική διεύρυνση. Επίσης, ε, διαπιστώσαμε συμμόρφωση με τους στόχους ε, στη δημιουργία των θεσμών. Δηλαδή ε, ε, προετοιμάζει τις χώρες αυτό το προενταξιακό μέσο για την ένταξή τους. Δημιουργούνται θεσμοί, εδραιώνεται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η οικονομική διακυβέρνηση. Διαπιστώσαμε στην έκθεσή σας και σημειώσαμε όπως και στην αξιολόγησή μας ότι εκφράζονται κάποιες ανησυχίες για ε, την έλλειψη αρνητική αιρεσιμότητα δηλαδή ρήτρε διακοπή αναστολή χρηματοδότηση. Και αυτό θα το λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό των νέων μέσων. Θέλετε ένα τέτοιο μηχανισμό, το σημειώνουμε και θέλουμε να συζητήσουμε την εφαρμογή του ε, επ' του στρατηγικού διαλόγου στις 22 Φεβρουαρίου. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του προενταξιακού μέσου έγιναν κάποιε πρόοδοι στη διοικητική και στην οικονομική διαχείριση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Τουρκίας. Διαπιστώσαμε και κάποιες δυσκολίες στην ε, απορρόφηση ε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την έμεση διαχείριση από τη δικαιούχο χώρα. Ε, όπως και με το μέσο της γειτονίας, ε, υπάρχει μεγάλη μόχλευση από το blending, από το συνδυασμό χρηματοδότησης με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Είναι πάρα πολύ πολύτιμη αυτή και μπορεί να κινητοποιήσει και ε, περαιτέρω χρηματοδότηση ε, από ιδιωτικούς πόρους. Προστιθέμενη αξία του πρωταξιακού μέσου, πολύ θετικό και εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλος δωρητής, ο πρώτος στις χώρες διεύρυνσης και έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα έτσι ώστε να υπάρξει απαραίτητο συντονισμός. Ακόμα και αν ο συντονισμός με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα όπως είναι το μέσο σταθερότητας και ε, ειρήνης ή κάποια άλλα χωράν βελτίωση. Πάντως γενικά υπάρχει ε, προστιθέμενη αξία. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φεράν. Περνάμε τώρα στον επόμενο μιλήτη. Κυρία Άνταμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω αναφορά στους προηγούμενους ε, ομιλητές και στην Κριστιαν. Τα μέσα που εφαρμόζονται από την εξωτερική πολιτική και που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ξεφεύγουν <coughs> από τα ορθόδοξα αυτά που συμβάλλουν στην δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ιδιαίτερα ελαστικά και γοργά βασίζονται σε συγκεκριμένες πολιτικές και οδηγούν σε μία γρήγορη ανταπόκριση που οδηγεί στην αλλαγή των πολιτικών προτεραιοτήτων. Είναι δηλαδή πολύ ε, ε, ευέλικτα και κινούνται σε ένα ευέλικτο περιβάλλον. Η ενδιάμεση αναθεώρηση συνέβαλε στο να είναι τα πλέον κατάλληλα αυτά τα μέσα και να δίνουν προστιθέμενη αξία σύμφωνη με τους στόχους που έχουν τεθεί. Αν κοιτάξουμε τα μέσα που συμβάλλουν στη σταθερότητα, θα διαπιστώσουμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος τους σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα προγράμματα, την ανοικοδόμηση της ε, ε, εμπιστοσύνη, ε, ειρηνευτικές διαδικασίες κτλ. Η ταχύτητα με την οποία κινούμε θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρόκειται για παράλληλα εργαλεία τα οποία συμπληρώνουν άλλα βασικά μέσα που ήδη υφίστανται. Και αυτό είναι κάτι που εξετάζουμε σε καθημερινή βάση έτσι ώστε να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τα μέσα αυτά και να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Αυτό είναι ένα σημείο όπου θα επιτείνουμε τις προτάσεις μας και τις παρεμβάσεις μας με βάση όσα μάθαμε από την ενδιάμεση αναθεώρηση. Να μιλήσουμε για το μέσο της εταιρική σχέσης. Δεν αποτελεί ένα συμβατικό μέσο συνεργασίας, αλλά για ένα μέσο που προφυλάσσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Το διεθνές πλαίσιο αναπτύσσεται και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό στρατηγικών προσεγγίσεων και προσαρμοστικότητας ε, στις, ε, συνθήκες που διαρκώς αλλάζουν. Σε μία σύσταση έγινε αναφορά σε αυτό ακριβώς το σημείο και θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε σε αυτά τα μέσα και που αφορά τις ε, υπηρεσίες εξωτερικές, εξωτερικής δράσης, ε, τα κράτη-μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους. Και πιστεύω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε μία ισορροπία μεταξύ του να εστιάζουμε σωστά και να είμαστε ελαστικοί. Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί και αυτό καθιστά αυτό το μέσον πάρα πολύ εμπέλικτο και του δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει τους στόχους του. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Αποστολή για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να πω ότι για μας είναι μια πραγματική ναυαρχίδα. Αυτό είναι ένα μέσο που εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση, αυτή η ελαστικότητα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των μέσων και στοιχεία που θα πρέπει να ενδυναμώσουμε στο μέλλον. Η κυρία Χακέη έθεσε το ερώτημα πώς συνεργαζόμαστε και πώς τα εφαρμόζουμε όλα αυτά. Μπορώ να πω ότι η συνεργασία μας με τις υπηρεσίες οδηγικές συνεργασίας είναι καθημερινή. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μας με τις άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. Και υπάρχουν άλλοι τρόποι συνεργασίας με άλλους εταίρους. Τώρα, να περάσουμε στο θέμα του ελέγχου. Ήδη αναφέρθηκε ότι υπάρχουν προοπτικές για περισσότερα μέσα στο μέλλον. Αυτά εξασφαλίζουν μια καλή, ένα καλό έλεγχο. Συγκεκριμένα μέσα μπορούν να γίνουν συγκεκριμένοι τρόποι παρέμβασης. Βεβαίως, για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξουν εξατομικευμένα μοντέλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε, ε, των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άνταμαν. Ο κύριος Βίλ. Thank you, Mr. Chair. Um, thank you Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η ομορφιά του να μιλάς τελευταίος είναι ότι σχεδόν όλα τα επιχειρήματα έχουν υποθεί, πράγμα που θα συντομεύσει και τη δική μου παρουσίαση, τουλάχιστον το ελπίζω. Θα επικεντρωθώ στο ADHR και να ε, θυμίσω λίγο περί τίνος πρόκειται. Ένα μικρό μέσο αυτό, συμπληρωματικό προς όλα τα υπόλοιπα και αφιερώνεται ιδιαίτερα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι μπορούμε παγκοσμίως να ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υποκαθιστά τίποτα, αλλά βοηθάει. Όπως σας είπα, έχει παγκόσμια κάλυψη, δηλαδή είμαστε παρόντες σχεδόν παντού. Δεν έχει περιορισμό ε, ως προς τους δικαιούχους και όρους. Κυρίως ε, συνεργαζόμαστε στη συντριπτική πλειονότητα με ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και όχι μόνο, μπορεί να είναι περιφερειακοί οργανισμοί οι διεθνείς οργανισμοί όπως το Γραφείο της Υπερδυσαρμοσίας στη Γενέβη και έχουμε το προνόμιο να εργαζόμαστε χωρίς να χρειαζόμαστε την έγκριση τη συγκατάθεση της τοπικής κυβέρνησης περιφερειακής ε, της εκάστοτε χώρας για να απτύξουμε τις δραστηριότητε μας. Στο βαθμό που το περιβάλλον βέβαια το επιτρέπει και μπορούν να εργάζονται οι ε, εταίροι μας. Η ΜΚΟ αυτή, ε, αυτό είναι ένας φυσικός περιορισμός, αλλά είναι ο μόνος. Όπως είπε και η Χίλντε, είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι, διότι έχουμε ειδικέ διαδικασίες ε, από τις οποίες επιφωλούμαστε ακριβώς για να δρούμε ταχύτατα όταν χρειάζεται. Και όντω το κάνουμε. Έχουμε πολλέ ιστορίε για υποστήριξη ατόμων, προσώπων ή οργανώσεων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ευέλικτα μπορούμε να τους υποστηρίζουμε σε επικίνδυνο περιβάλλον. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε και με φυσικά πρόσωπα. Δεν χρειάζεται κάποιο να, είναι, να έχει καταχωρηθεί κάπου, να είναι μια οργάνωση, να είναι νομικό πρόσωπο, όταν ε, υπάρχουν δυσκολίες και κίνδυνοι. Το 60% της δράσης μας Ε, είναι αντικείμενο διαχείριση επιτόπου, που είναι η καλύτερη διαχείριση γιατί γνωρίζουν ε, την εκάστοτε κατάσταση που επικρατεί οι ενδιαφερόμενοι. Αυτά για να σας δώσω το πλαίσιο. Ε, για την ενδιάμεση θεώρηση. Είναι αποτελεσματικό αυτό το μέσο. Μάλιστα. Από την έγκρισή του, ιδιαίτερα στα πλαίσια των προβλημάτων που έχουν οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους οποίους βοηθούμε παγκοσμίως, εγγράφεται στην Ατζέντα 2030 και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, τα στοιχεία της ε, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα, θα πρέπει βεβαίως να ενσωματωθούν εκεί. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του μέσου, πέρα από τη σκοτιμότητα, όλες οι δράσεις έχουν ειδικού στόχους, άρα θεωρήθηκε το μέσο αποτελεσματικό μέχρι στιγμής υποστηρίζει βασικές προτεραιότητες τώρα όπως η μετανάστευση, η ειρήνη, η ασφάλεια όχι με την αμεσότητα που θα θέλαμε ίσως οι αποστολές παρατηρήσεις εκλογών είναι αποτελεσματικές και προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το μέσο αποδείχτηκε και θεωρήθηκε αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο υπάρχουν στοιχεία που λέγουν ότι είμαστε και εκεί αποτελεσματικοί Έχουμε σώσει τη ζωή ε, αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές περιπτώσεις. Τι αντίκτυπο έχουμε και τι γεωγραφική διασπορά σε σχέση και με τον περιορισμένο προπολογισμό. Έχουν γίνει προτάσει να εστιάζουμε περισσότερο σε χώρε που γνωρίζουν κρίση. Βέβαια, πάντα από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κατεπίγουσε καταστάσει, σε δύσκολε περιπτώσει. Ε, αυτό είναι πάντα πρόκληση όπου κινδυνεύουν περισσότερο δηλαδή αυτοί οι ακτιβιστές και να κοιτάξουμε τι γίνεται με τους δημοσιογράφους ή κάποιες ε, ομάδες που γίνονται στόχος ε, η ΛΟΑΔ και άλλες ομάδες που στοχοποιούνται συχνά. Λοιπόν, είναι καλή η ροή, ε, η εκταμίευση των χρημάτων, είναι αποτελεσματικό το ταμείο, πιάνουν τόπο τα χρήματα, ε, γίνεται καλή χρήση της ε, ενότητας ε, για την ευελιξία. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε φυσικά πάντα την κατάσταση. Τα φυσικά πρόσωπα είναι κάτι στο οποίο επιμένω να απευθυνόμαστε περισσότερο σε φυσικά πρόσωπα. Βεβαίως οι δείκτες να βελτιωθούν. Τώρα να θεωρούμε όλο το σύστημα των δικτών, όχι μόνο τους δικούς μας για το συγκεκριμένο μέσο και αυτό θα συνεισφέρει στην κατεύθυνση που είπε και η συγκήτρια κυρία Σχάκε για το Κοινοβούλιο και το δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συμφωνούμε απολύτω. Έχουμε προβλήματα με τις προκηρύξεις των διαγωνισμών. Καμιά φορά είναι βαριές διαδικασίες, γραφειοκρατικές, χρειάζονται πολλές άνθρωπο και εμείς ε, υποφέρουμε από τη διαχείριση σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό. Συμπληρωματικότητα, όπως σας είπα, είναι μοναδική έρχεται να καλύψει κενά σε κάποιες δύσκολες ε, καταστάσεις όπου άλλοι δωρητές ή κάποια κράτη-μέλη αποχωρούν και δεν ασχολούνται με το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την πολιτική μόχλευση, μπορούμε να ενισχύσουμε τους μεταρρυθμιστές και τους αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκάστοτε χώρα. Και τέλος, για τις συστάσεις, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μακρηγορώ, θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στους αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον πρώτο στόχο, σε δύσκολες καταστάσεις, όπως σας είπα. Υπάρχει πραγματικά ε, ανάγκη και ζήτηση και θα πρέπει να προσανατολιστούμε περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε να υποστηρίξουμε και τα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων και τα κοινοβούλια, γιατί και αυτό είναι στοιχείο Δημοκρατία. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ, γιατί αλλιώ θα με ακριβώσω πάρα πολύ και δεν θα το ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βίλ. Ακούσαμε λοιπόν τους τέσσερις ομιλητές από τα ευρωπαϊκά όργανα. Τώρα περνάμε στους φιλοξενούμενους. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σέρεφ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόσκλησή της. Αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να κοιτάξω προς το μέλλον πώς ε, θα μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η ελαστικότητα, εσωτερικές και εξωτερικές ε, πολιτικές και ε, εξορθολογισμός στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτής της συζήτησης θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε από πάνω προς τα κάτω και όχι ε, από κάτω προς τα πάνω και όχι μόνο από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε αλλάξει πάρα πολύ Αυτό είναι κάτι που καθίσταται σαφές στην διάμεση αναθεώρηση αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που έχουμε μάθει να, ε, να κάνουμε. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής είναι ότι τα μέσα είναι κατάλληλα για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αναρωτιέμαι αν αυτή είναι μια πολιτική απόφαση και ότι θα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό το λόγο δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα <clears throat> Τώρα, μόνο ότι υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν και νέες ευκαιρίες. Έχουμε μια γενική στρατηγική, έχουμε το χρονοδιάγραμμα το 2030, αυτά που δεν είχαμε πριν από τη διαπραγμάτευση του τελευταίου πολιετούς πλαισίου. Έχουμε λοιπόν ένα νέο χρονοδιάγραμμα, ένα σαφέστερο χρονοδιάγραμμα από ό,τι στο παρελθόν τα εξωτερικές υποθέσεις έχουν επανέλθει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν σημαντικές διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές. Ένα από τους προβληματισμούς που έχουμε έχει σχέση με το ότι θα μπορούσε να εκφυλιστεί η συζήτηση σε θέματα πρακτικά. Πόσα χρήματα θα χρειαστούν για την πίστοση Α, για την πίστοση Β, για... και δεν θα υπάρξει μια στρατηγική σημασία για τα τι και τα πώς. Οι βασικές προκλήσεις τώρα. Η πρώτη είναι η ευελιξία και αυτό εμφανίζεται σε κάθε είδους συζήτηση. Ενδεχομένω μερικοί από εσά αναρωτιούνται γιατί τη μία φορά βλέπω μία πάπια, την άλλη φορά βλέπω ένα κουνέλι κοιτάζοντας την ίδια εικόνα. Η ελαστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορούσαμε να την ε, διαχειριστούμε. Πολλά έχουν σχέση με τη μόχλευση ε, νέων πόρων ή τη δημιουργία, ε, την συνεργασία με άλλους εταίρους. Επίσης είμαστε διατεθειμένοι να παρετηθούμε ενό μέρους της επιρροής μας στο όνομα περισσότερης ελαστικότητας ή να βρούμε φιέστερους τρόπους για να εξασφαλίσουμε την ευελιξία και να υπάρχει παράλληλα και χρηστή διαχείριση. Η ευελιξία δεν είναι κατά ανάγκη ένα πολύ γερό θεμέλιο. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Η ευελιξία όμως είναι ο όρος που επανέρχεται πάρα πολύ συχνά. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία, τίθεται το θέμα των αξιών προς τα συμφέροντα ως αξιολογητές γίνεται μια συχνή αναφορά στον όρο προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα και να μην ε, χαθούν όλα αυτά ε, λαμβάνοντας υπόψη εθνικά συμφέροντα. Η ευελιξία λοιπόν δεν θα πρέπει να υπονομεύσει όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά το, τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα, εμείς δεν ορίζουμε ένα προπολογισμό γιατί το 2050. Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και το θέμα είναι το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα. Είναι αυτό που μετράει. Νομίζω ότι τα εργαλεία της συνεργασίας είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να προφυλάξουμε για την εξωτερική χρηματοδότηση και να μην χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια μόνο για σκοπούς που αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αξίες και συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί ποιες είναι οι αξίες της και αυτό ισχύει και για αυτό που συμβαίνει μέσα στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής. Άλλες χώρες έχουν άλλους εταίρους, άλλες αξίες και υπάρχουν τομείς που αφιλού, απειλούνται πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Θα πρέπει να δει κανείς ποιο είναι το συμφέρον του και από την άλλη πλευρά ποιες είναι οι αξίες του. Και πάρα πολλές φορές ασκούνται πιέσεις στις αντιπροσωπείες οι οποίες θα πρέπει να καταβάλουν μια προσπάθεια να συγκεράσουν και τα δύο. Ο εξορθολογισμός. Ένα από τα θέματα που τίθεται συχνά είναι η δημιουργία ενός ενιαίου μέσου. Δεν θα υπάρξει ένα μέσο που θα μπορούσε να συνδυάσει τα πάντα σε ένα. Τι Τίθεται λοιπόν το ερώτημα τι θα κρατήσουμε, τι θα αφήσουμε απ' έξω. Ένα ενιαίο μέσο θα μπορούσε να βοηθήσει τον εξορθολογισμό αλλά βεβαίω ε, δεν είναι το μαγικό ραβδί για την έλλειψη πολιτικών κατευθύνσεων ή για στρατηγικό έλλειμμα. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Ποιο θα είναι το όλο αφήγημα που θα μπορούσε να αιτιολογήσει ένα ενιαίο μέσο. Τι είναι, είναι η παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη, θα μπορούσε να υπάρχει ένα μέσο για την Αφρική ή θα υπάρχει ένα και μοναδικό μέσο παγκοσμίω. Ποιες είναι οι διάφορες δομές ε, της ε, διαχείρισης, τι συμβαίνει με τη λογοδοσία και αν υπάρχει ένα και μοναδικό ε, μέσο με διάφορα κεφάλαια και διάφορα, με διάφορα κονδύλια Μήπως επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα που ήδη υπάρχει. Το θέμα είναι τι θα συμπεριλάβουμε εδώ από το τρέχον μέσο. Και τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Συμπεράσματα. Υπάρχει ανάγκη για στρατηγική αντιμετώπιση, αλλά ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Τι, για τι είδους ευελιξία μιλάμε, για τι είδους αρχιτεκτονική, για τι είδους ε, κονδύλια. Ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, όπως είπαμε. Πολύ σωστά αυτή είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία θα είναι κρίμα στο τέλος του, της διαδικασίας του πολιετούς πλαισίου να έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο αλλά από τη μία πλευρά, από την άλλη οι εταίροι να είναι απογοητευμένοι και να θεωρούν ότι αυτό το τελικό προϊόν δεν αντικατοπτρίζει τις δικές τους ανησυχίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σωστές διαβουλεύσεις με τους εταίρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ιωαννίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Όπως γνωρίζετε, η εκ των υστέρων αξιολόγηση γίνεται από την ε, αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Έρευνας. Έχετε ήδη λάβει την αρχική διατύπωση την οποία είχα προτείνει για την Επιτροπή ΑΦΕΤ προσπαθώντας να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε τους εισηγητές που εργάζονται σε αυτό. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάκε και την Γραμματεία της Επιτροπής για την εξαιρετική του συνεργασία. Η μελέτη την οποία λάβατε σήμερα αξιολογεί κάθε μέσο ξεχωριστά Προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε στο σύνολο των εξωτερικών μέσων χρηματοδότησης και υπογραμμίζουμε παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μετά από την αρχιτεκτονική που θα ακολουθήσει τα μέσα αυτά μετά το 2020. Υπάρχει επίσης και ένα έγγραφο εμπειρογνωμοσύνης ε, το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένα μέσα στήριξης όπως αυτό για την Τουρκία, την Ουκρανία και την Αίγυπτο. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Λεφλέρ γιατί νομίζω ότι κάποια από τα σημεία τα οποία εμείς συστήνουμε περιλαμβάνονται ήδη σε αυτά τα οποία μας είπε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και αυτό το βρίσκω θετικό. Θα ξεκινήσω από εκεί που μπορεί να διαφωνούμε περισσότερο. Όταν επιλέγουμε την διαδικασία της απλοποίησης έτσι ώστε να προστατευθούμε από την υπεραπλούστευση. Πράγματι εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά σε όλα τα μέσα ξεχωριστά. Η βασική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε και την οποία είδαμε και στην εφαρμογή του μέσου αυτού ε, έχει σχέση με τους ε, δεσμούς οι οποίοι δημιουργούνται από το πέρασμα ε, από τη μία φάση στην επόμενη. Είναι κάτι το οποίο έχει, θα έλεγα, ισχύει για όλα τα μέσα και όχι μόνο για ένα συγκεκριμένο. Η συμπληρωματικότητα λοιπόν είναι ο στόχος και το λεγόμενο streamlining και βλέπουμε ότι τα μέσα αυτά έχουν σαν στόχο να καλύψουν τις ανάγκες χωρών με τις οποίες έχουμε προχωρήσει σε επίπεδο περιφερειακής συνεργασίας, αντιμετωπίζοντας όμως και αναγνωρίζοντας τα ειδικά τους περιφερειακά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό όταν μιλάμε για χώρες εύθραστες ή για χώρες μεσαίου επίπεδου, θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα συγκέντρωσης ορισμένων μέσων εδώ στις Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα κάποια άλλα μέσα να παραμένουν ανεξάρτητα. Να είμαστε επίσης ε, βέβαιοι ότι ένα μεγαλύτερο μέσο δεν σημαίνει υποχρεωτικά επιβαρημένη γραφειοκρατία. Δεν θα πρέπει εμείς όταν προσπαθούμε να πετύχουμε την ευελιξία να την δυσκολεύουμε στην ουσία. Ένα δεύτερο θέμα είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την συνέχεια και την βιωσιμότητα των μέσων αυτών. Υπάρχουν ένα από τα όρια που έχει η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι ότι έχει συγκεκριμένα μέσα προγράμματα και βάσεις στη διάθεση. Οπότε δεν είναι γενικής εφαρμογής και δεν πετυχαίνει το σύνολο των στόχων. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά τις καλές προθέσεις που υπάρχουν για την προσπάθεια της ενίσχυσης της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, του εκδημοκρατισμού και του σεβασμού του κράτους δικαίου, τελικά εμείς πιέζουμε περισσότερο όχι τόσο για τη δημοκρατία αλλά για τη σταθερότητα. Ένα τρίτο θέμα είναι η διευκόλυνση της ευελιξίας. Μιας και μιλάμε για χρηματοδοτικά μέσα, θα αναφερθώ στη ρευστότητα που διασφαλίσουν οι πιστώσεις αυτές. Όπως είδαμε και στο παρόν πολιετές δημοσιονομικό το επίπεδο ευελιξίας εξαρτάται από τα διαθέσιμα ανώτατα όρια. Τα χαμηλά ανώτατα όρια τα οποία ισχύουν σήμερα έχουν πραγματικά οδηγήσει τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς να λειτουργούν στο όριο καλύπτοντας πολλές από τις ανάγκες κάλυψης ε, χωρίς στήριξη. Πρέπει λοιπόν τα χρηματοδοτικά μέσα να έχουν την δυνατότητα να μετακινούν πιστώσεις εάν αυτό χρειάζεται για να καλύπτουν ακριβώς και κάποιες νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε νέες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει επίσης και η συνεκτικότητα να συνοδεύει την ευελιξία. Ε, πράγματι υπάρχουν νέα μέσα επικοινωνίας, ιδιαίτερα στον τομέα της μετανάστευσης με τα λεγόμενα νέου τύπου καταπιστεύματα. Αλλά το αποτέλεσμα μέχρι τώρα της προσπάθειας μας είναι ενδιάμεσης ποιότητας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε το εξής ερώτημα σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να πετυχαίνουμε αποτελέσματα ιδιαίτερα όταν οι κυβερνήσεις οι οποίες είναι αυτές που ωφελούνται ε, δεν ε, συμφωνούν με την αιρεσιμότητα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Θα πρέπει εδώ να ενισχύσουμε λοιπόν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, τις διαιτητικές διαδικασίες και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε νέους κανόνες στα χρηματοδοτικά μέσα που να απαιτούν στους εκπροσώπους από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να είναι σε άμεση επαφή με τις κυβερνήσεις δικαιούχους θα έλεγα των ε, προγραμμάτων αυτών. Να στηρίξουμε επίσης και την κοινωνία των πολιτών, να έχουμε σχέσεις και δεσμούς όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση πολλών από τις χώρες αυτές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να δημιουργήσουμε επίσης διαφορετικές κατηγορίες χρηματοδότησης της κοινωνίας των πολιτών. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας μέσος όρος, ένας μηχανισμός ο οποίος να είναι ικανός να καλύψει όλες τις ανάγκες. και κυρίως όχι τις ανάγκες που να συνδέονται μόνο με την κυβέρνηση κάθε φορά. Τώρα στρατηγική και δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται στόχοι οι οποίοι να είναι πιο συγκεκριμένοι και θα πρέπει επίσης να υπάρχουν εταιρικέ σχέσεις με πολλαπλούς παραλήπτες έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και τον ρόλο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίζουν κομβικό ρόλο για να εντοπίζουν ακριβώς ποιοτικά τουλάχιστον τους συνομιλητές μας επιτόπου. Να μην λειτουργούμε μόνο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δυτικότροπες, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε ποιες είναι αυτές που πολλές φορές δεν είναι προφανείς, οι οποίες όμως είναι αντιπροσωπευτικές. Και τέλος, να ενισχύσουμε την στρατηγική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικοινωνίας. Εδώ θα ήθελα να ζητήσω περισσότερη στήριξη ε, για επικοινωνία με τα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης, περισσότερη χρηματοδότηση έτσι ώστε η πολιτική μας να γίνεται κατανοητή στις χώρες δικαιούχους και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο όλους τους εμπλεκομένους και τις επαφές με εμπλεκομένους που έχουμε σε κάθε χώρα. και μέσω των δικτύων των πρεσβειών και μέσω των αντιπροσωπιών και των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανώσεων. Έτσι θα μπορέσουμε λοιπόν να πάρουμε μαθήματα από τις τοπικές εμπειρίες και να διευκελύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Πραγματικά δεν έχουμε χρόνο κυρία Ιωνίδη στην διάθεσή μας και έχουμε άλλους δύο μιλητές και μετά θα στραφούμε στα μέλη. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι να κάνετε ερωτήσεις, να τις κάνετε παρακαλώ σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Το βασικό μου συμπέρασμα για την υποστήριξη στην κοινωνία των πολιτών ε, είναι ότι έχει αυξηθεί και έχουν αυξηθεί και τα ποσά με τρόπο πιο ευέλικτο χορηγεί τη βοήθεια και πιο προσανατολισμένο στις ε, στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές. Είναι πολύ χρήσιμη η εργασία μας. Προστατεύουμε ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις που απειλούνται από καθεστώτα και κυβερνήσεις. Σε πολλές χώρες έχει επιθυνωθεί η κατάσταση της κοινωνίας πολιτών και η δομή και η διάρθρωσή τους αλλάζει με δραματικό τρόπο. Στον τομέα αυτό τα γεγονότα στον πραγματικό κόσμο μετά την Ευρωπαϊκή και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ζητούν αναθεώρηση των χρηματοδοτικών μέσων. Η Αίγυπτος και η Τουρκία δύσκολες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει εφευρετικότητα και έχει ε, βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών, ε, αλλά γενικότερα δεν έχει προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκρούσει τις επιθέσεις που δέχεται η κοινωνία των πολιτών. Στην Ουκρανία ενισχύουμε την κοινωνία των πολιτών και αυτό βοηθάει τις μεταρρυθμίσεις σε πολύ σημαντικό τρόπο αλλά και πάλι υπάρχουν προβλήματα, ελλείψεις, ανισορροπίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να βελτιωθεί για το μέλλον. Αν υπάρξει ένα μοναδικό μέσο ε, θα ε, βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών, αλλά εδώ υπάρχουν διάφορες ευαισθησίες όπου χρειάζονται διάφοροι τρόποι υποστήριξη και διάφοροι κανόνε. Ε, αντίστοιχα, αν υπάρξει ένα και μόνο μέσο για την κοινωνία των πολιτών μπορεί να περιπλακεί η κατάσταση πάρα πολύ. Τι προτείνω λοιπόν, να διατηρηθεί η παρούσα δομή, αλλά κάπως να συντονιστεί ε, η υποστήριξη κοινωνίας των πολιτών για να έχουμε μια γενικότερη εικόνα το πώς ε, είναι η κοινωνία των πολιτών και πώς ε, χρειάζεται να ενισχύεται. Πολλές φορές είναι συγκεχημένη η εικόνα για το τι είναι η κοινωνία των πολιτών ε, σε κάθε χώρα, τι κάνει και ποιοι είναι στατηγικοί στόχοι. Βασικός στόχος για μένα εδώ ποιος είναι. Καλύτερη σύνδεση της υποστήριξης της ε, κοινωνίας των πολιτών με άλλη μορφή βοήθειας για τις μεταρρυθμίσεις κλπ. Αυτό λείπει συνήθως στις τρίτες χώρες. Ενισχύουμε διάφορους τομείς μεταρρυθμίσεις με τρόπο αποσπασματικό και όχι ενιαίο. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε ο Ζαν Λουί υπάρχει χώρο για περισσότερη ευελιξία και λόγο. Αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή η βασική προτεραιότητα ούτε πανάκια στην κοινωνία των πολιτών αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Δεν χρειάζεται καμιά ανακατασκευή της αρχιτεκτονικής. Η πολιτική βούληση είναι αυτή που λείπει από τα κράτη-μέλη να βάλει ως προτεραιότητα ε, την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Ε, τώρα, βασική προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη που έχει τα τελευταία χρόνια επιδεινωθεί είναι να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Έχει επιδεινωθεί πολύ το πρόβλημα και είναι πολύ πιο συστηματικό από την εποχή που σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά τα μέσα. Χρειάζονται επικαιροποίηση, ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικός στόχος πρέπει να αλλάξουν και οι διαδικασίε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει καλύτερα τι οργανώσει, των πολιτών, μάλλον τη κοινωνία των πολιτών που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολε καταστάσει. Ε, δύο τελευταία για να κλείσω. Ακριβώ επειδή αλλάζει η κοινωνία των πολιτών ανά τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα για να στηρίξει νέου ακτιβιστέ και νέε οργανώσει έχει γίνει κάποια προσαρμογή, έχουν εξελιχθεί κάπως τα μέσα, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη αλλαγή. Και το τελευταίο, θεωρητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη στην υποστήριξη ε, της κοινωνίας των πολιτών σε ένα πλαίσιο γενικότερο στόχο, Αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ καλούς μηχανισμούς για να το ελέγχουμε αυτό αν γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες, κάποια κριτήρια που είναι τόσο γενικά που οποιαδήποτε στήριξη της κοινωνίας των πολιτών να θεωρείται ότι ε, εντάσσεται στο στόχο. Εδώ χρειάζεται πολύ περισσότερη ακρίβεια και καλύτερη ευθυγράμμιση με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να εστιάσει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση στο χαρακτήρα της ασφάλειας ε, γιατί αν το κάνει αυτό θα χάσει πολλά από τα καλά ε, σημεία που υπάρχουν σήμερα για την υποστήριξη κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat> Περνάμε στον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Ζιβανίδη. Την κυρία Ζιβανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πολλές ε, οργανώσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και ασχολούνται με το θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε μια χρηματοδότηση από την PSC και άλλες οργανώσεις μέλη και θα ήθελα να αναφερθώ στην ICSP και θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Πιστεύω ότι έγινε μια αναφορά στον κόσμο που αλλάζει και στην κρίση που καλούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε και στο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. αξία της Ευρωπαϊκής Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές. Θα μπορούσα να αναφερθώ στα θέματα ασφαλείας, στα θέματα άμυνας, Εμείς καταβάλουμε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε θέματα ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι όμως που θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα ε, οδηγήσει αυτόματα στην επίτευξη ειρήνης. Στην έκθεση της, ε, στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει βασικά θέματα ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι είναι το μοναδικό εξωτερικό εργαλείο που ευστιάζεται στην αποφυγή των σειράξεων και που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τις αξίες της. Σε αυτή την άποψη τη συμμερίζονται οργανώσεις ε, δικές μας αλλά και εξωτερικές οργανώσεις που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Επίσης ε, γνωρίζουμε ότι οι αναφορές στην ΕΣΤΕΠΗ αναφέρονται στην ασφάλεια στα σύνορα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας ενιαίος τομέας που συμβάλλει στην ε, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια στα σύνορα, αλλά που είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικά. Μιλώντας για την ειρήνη και την ασφάλεια, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για αυτά τα θέματα, ε, θέματα που αφορούν τα θύματα ένοπλων συγκρούσεων, την ειρήνη σε χώρες όπου λαμβάνουν χώρα αυτά τα πάνθρωπα <clears throat> γεγονότα, την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και την... Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι τα θέματα που θα πρέπει να μας ασχολούν η έγκαιρη, η προειδοποίηση. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα ε, θετικά στοιχεία που αφορούν το μέσο συμβουλή στη σταθερότητα και την ειρήνη, το ICSP. Θα πρέπει επίσης ε, να μας απασχολήσει, το πώς θα εφαρμοστεί η το πρόγραμμα που αφορά τη συμβολή των γυναικών στην ειρήνη. Υπάρχει προσωπικό σε επίπεδο περιφερειακό και σε επίπεδο Βρυξελών που φροντίζει, που ξέρει πόσο θα πρέπει να κινηθεί σε αυτό το τομέα. Και ξέρω ότι υπάρχουν αυτοί που τα καταλαβαίνουν καλά και που χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα. Στο Αφγανιστάν όμως ε, για παράδειγμα ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν εννοούμε ακριβώς ε, το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας την ίδια ορολογία. Δεν υπάρχουν μέσα τα οποία είναι κατάλληλα για κάθε περίσταση. Δεν θα μιλήσω για θέματα που έχουν ήδη θυγεί. Είναι σημαντικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διατηρηθεί το μέσο συμβολή στη σταθερότητα και την ειρήνη. Νομίζω ότι το θέμα της ευελιξίας παραμένει και αυτό ένα κεντρικό θέμα. Υπάρχουν ε, πολλά ε, ερωτήματα εδώ. Είναι σαν ένα ντουλάπι με πολλά σιτάρια που ανήκουμε κάθε φορά και το σίγουρο είναι ότι ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Το ICSP, το μέσο συμπολής, είναι το πιο ευέλικτο μέσο και η πρόληψη των σειράξεων αποτελούν μέρος αυτού του μέσου. Αυτό καθίσατε σαφές στην γενική στρατηγική φιλοδοξίες μας, ε, δηλαδή σε αυτό το τομέα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Η άποψη της Επιτροπής για την έκθεση ζητάει να διατηρηθούν ξεχωριστά μέσα με ξεχωριστούς ρόλους. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της και να προετοιμάσει τα μέσα για το επόμενο πολιετές πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ σε όλους τους ομιλητές και ζητώ συγγνώμη που σας πίεσα. Οι συνάδελφοι τώρα δεν ξέρω αν έχουν να θέσουν ερωτήσεις. Ο κύριος Κουκάν. Δεν έχω ακριβώς ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να κάνω αρκετές παρατηρήσεις Εγώ ήμουν εισηγητής για τα θέματα γειτονίας. Ενθυμούμε ότι πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλές απαιτήσει από πλευράς ε, κάναμε πολλές παραχωρήσεις από πλευράς της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και υποχωρήσαμε στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήταν λάθος αυτό. Από ό,τι φαίνεται το Κοινοβούλιο έχει ελάχιστο έλεγχο σε σχέση με τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα και έχει επίσης πολύ μικρή πολιτική παρέμβαση. Και ανησυχώ και μου κάνει εντύπωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν μπορούν να μας δώσουν μια απλή αξιολόγηση της λειτουργίας των μέσων αυτών δεν βρήκα τις απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέσα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή τους κτλ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είτε είναι πάρα πολύ γενικού τύπου ε, και γενικά θολές στην κατανόησή τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση γύρω από αυτό. Ακόμα και η βασική αρχή more for more, η οποία είχε συζητηθεί πάρα πολύ, πώς εφαρμόστηκε. Είμαι περίεργος. Ήταν αποτελεσματικό μέσω στις σχέσεις μας με τις υπόλοιπες χώρες ή όχι. Δεν πήρα καμία απάντηση. Δεν θέλω να μακρηγορώ, αλλά θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για την αρχιτεκτονική των μέσων αυτών. Από τη μία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι τα μέσα αυτά είναι κατάλληλα και δεν απαιτούνται νομοθετικού τύπου ε, αλλαγές και τροποποιήσεις ή ε, ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Ακούω όμως από συναδέλφους και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής της αρχιτεκτονικής. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί χρειάζεται να αλλάξουν τα μέσα αυτά. Εγώ δεν είμαι κατά φυσικά των αλλαγών εφόσον ενισχύσουν τις εξωτερικές μας πολιτικές δραστηριότητες και προτεραιότητες. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι αλλαγές αυτές προτείνονται μετά από κάποιες διοργανικές επαφές και συζητήσεις και αυτό είναι λάθος και με βρίσκει να διαφωνώ. Λοιπόν, τελειώνοντα για το μέλλον θα θέλω να πω ότι απαιτούνται μέσα τα οποία πράγματι να είναι αρκετά ευέλικτα. Υπάρχουν πάρα πολλέ εξελίξεις ε, ουσιαστικέ στον κόσμο, μετανάστευση, σχέσεις με Ρωσία κτλ. Και τα μέσα θα πρέπει να είναι λοιπόν αρκετά ευέλικτα έτσι ώστε να προσαρμόσουν την κατάσταση στις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να επηρεάζει περισσότερο από ό,τι σήμερα και να συναποφασίζει στη χάραξη των πολιτικών. Ευχαριστώ. Κριστέα, να ευχαριστήσω, ε, να στηρίξω αυτά τα οποία είπε ο κ. Κουκάνη. Ήμουν σκιώδης εισηγητής για το θέμα αυτό και για τα προενταξιακά μέσα εδώ και δύο-τρία χρόνια. Οι εμπειρίες από την τροποποίηση και την απλούστευση της αρχιτεκτονικής αυτών των μέσων ε, είναι πραγματικά μια σαφής ανάγκη και υπάρχουν αρκετές ε, προτάσεις, υπάρχουν τρία τουλάχιστον σενάρια μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως κάποιες αλλαγές ε, τέτοιου είδους να φαίνονται τεχνικές, είναι όμως βαθιά πολιτικές. Νομίζω ότι θα φέρουν στην επιφάνεια όλες ε, όλες τις καταστάσεις σύγκρουσης ε, ισχύω που μπορεί να σοφούν σε διάφορες χώρες και στα ευρωπαϊκά όργανα. Τώρα για τις μελλοντικέ εκθέσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική γειτονίας είναι σαφές ότι δεν μπορούμε πια να αγνοούμε τις διαφορές και τις διαφωνίες που έχουμε σε σχέση με τις εξελίξεις Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία και οι τρεις αυτές χώρες ε, πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να αναλάβουν πολιτικές υποχρεώσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή τους πορεία και γι' αυτό απαιτείται να υπάρξει ένα πολιτικό όραμα για αυτούς οι οποίοι στρέφουν τις χώρες αυτές προς την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ζητάμε λοιπόν τα ειδικά ταμεία για τις τρεις αυτές χώρες να μην ακολουθήσει τις, την πορεία την οποία ακολούθησε μέχρι τώρα. Πέρυσι στη συνάντηση κορυφής δεν έγινε καμία αναφορά στις προτάσεις τις οποίες έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτές τις τρεις χώρες, οι οποίες μετά το 2020 είναι υποψήφιες προσένταξη χώρες, αν τις βάζουμε στο ίδιο καλάθι με όλες τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ πολύ για Στρεβίτσιους. Ευχαριστώ Μαρίσα, ευχαριστώ και για την ε, γραπτή σου πρόταση η οποία είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για το μέλλον των ε, εξωτερικών αυτών μέσων. Ευχαριστώ επίσης και όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει πράγματι να αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής και να είναι σύμβατες με τις στρατηγικές τις οποίες έχουμε ήδη ε, και αρκετές θα έλεγα στην Ένωση. Το θέμα είναι πώς θα συντονιστούν καλύτερα, πώς θα τις καθοδηγήσουμε τις πολιτικές αυτές. Αυτή είναι η δυσκολία σήμερα και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν την διαχείριση των πολιτικών αυτών σε πολιτικό επίπεδο να την ενισχύσουμε. Και αυτό θα γίνει μέσα και από τη συμμετοχή των υπεύθυνων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πώς μπορούμε να μειώσουμε επίσης την περίοδο ανάμεσα στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή του μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα μερικές φορές στους δικαιούχους, στις ΜΚΟ και τα λοιπά και μερικές φορές το χρονικό διάστημα το οποίο διαμεσολαβεί δεν μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε επίγουσες ανάγκες. Αρτιότερες ε, πολιτικές στον τομέα της επικοινωνίας είναι κάτι το οποίο μας χρειάζεται έτσι ώστε να αξιγούμε στους εταίρους μας και τους συνεργάτες το τι ακριβώς κάνουμε. Εφαρμογή και μέσα διαθέσιμα. Ε, νομίζω ότι η έλλειψη ερεσιμότητας μπορεί να οδηγήσει και σε αποτυχίες ακόμα και η μικροοικονομική αν θέλετε βοήθεια ε, πολλές φορές ε, πρέπει να συνοδεύεται από αιρεσιμότητες πολιτικού τύπου. Είναι κάτι το οποίο απαιτείται, δεν είναι ένα δώρο χωρίς προϋποθέσεις. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η αρχή της αιρεσιμότητας και να ενισχυθεί. Και δεν μιλάμε μόνο για το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τα κράτη-μέλη, τα οποία χρησιμοποιούν δικά τους μέσα βοήθειας. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα μέσα αυτά να συνδυάσουμε καλύτερα τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ευρωπαϊκών μέσων. Ευχαριστώ κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, περιμένω λίγο να βάλετε τα ακουστικά σας. Ε, η θέση της δικής μου πολιτικής ομάδας είναι πολύ επικριτική. Καταρχήν, έχουμε επιφυλάξεις απέναντι στο μέσο σταθερότητας και ειρήνης ιδιαίτερα στη στήριξη στρατιωτικών ε, φορέων. Αλλά δεν θέλω να πω τίποτα σχετικά με αυτό. Εκφράζω τις καταρχήν επιφυλάξεις μου, της ομάδας μου. Για τον έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό και τη συναπόφαση θέλω να μιλήσω. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, έχω κάποια εμπειρία μερικών ετών ε, στις ομάδες εργασίας και πρέπει να σας πω ότι σε αυτές τις ομάδες εργασίας που κάνουν την αξιολόγηση υποτίθεται πώς να το πω, θα σας φανεί λίγο σκληρό, αλλά πώς να το πω διαφορετικά, είναι σκέτη φάρσα αυτές τις ομάδες εργασίας. Ποια αξιολόγηση. Όλο ακούμε ότι ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες ε, να τον δούμε όλα στο διαβολάκο αυτόν που είναι στι λεπτομέρειε. Αν δεν μπούμε ποτέ στι λεπτομέρειε, δεν θα το γνωρίσουμε. Και μετά ακούμε δηλώσει τύπου, αυτά που λέει η κυρία Χάρτεμαν, στην Τινησία η μακροοικονομική σταθερότητα βελτιώθηκε. Μυστήριο πράγμα, ο κόσμος διαδηλώνει λόγω της μακροοικονομικής αστάθειας που τους έχει πλήξει. Ακόμα και τέτοια συγκεκριμένα που μας λέτε για συγκεκριμένες χώρες δεν στηρίζονται πουθενά, είναι κούφια λόγια. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες δυνατότητες ελέγχου, συμμετοχής, αξιολόγησης με δική μας συμμετοχή. Έχω και κάποια ερωτήματα πάλι αρχής. Η δική μου πολιτική ομάδα ανέκαθεν αγωνιζόταν για το μέσο σταθερότητας ε, να υπάρχουν και εκεί κατεξιολόδότηση πράξης που δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Αλλά υπάρχουν άλλα μέσα που δίνουν αυτή τη δυνατότητα των κατεξιολόδότηση πράξεων και τώρα αυτά τα παραγνωρίζετε θα πρέπει κανείς να έχει την ενέργεια και το κουράγιο ενός ερευνητικού δημοσιογράφου για να πάει να ψάξει τι γίνεται με το μέσο ας πούμε της γειτονίας που δίνονται κονδύλια για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κανονικά θα έπρεπε να αλλάξει η περιγραφή ε, του μέσου και κατεξοδότηση πράξης να ακολουθήσουν τίποτα από όλα αυτά παίρνουν τα λεφτά από το πρωταξιακό μέσο, από τη γειτονία μάλλον και το δίνουν στην Τουρκία. Ο, κατά το δοκούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος να πω ότι έχω μεγάλες επιφυλάξεις και αρχής πάλι σχετικά με την σχέση του προγραμματιζόμενου και μη προγραμματιζόμενου τμήματος ε, του Ταμείου και του μέσου που και αυτό διεφεύγει το έλεγχο. Περισσότερη ευελιξία πρεσβεύεται όλοι. Και πώς να έρθει όλος να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο όταν θέλετε περισσότερη ευελιξία. Αυτά. Ευχαριστώ. τον Thank Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να ακουστούν οι απόψεις των διαφόρων πλευρών και πιστεύω το νόημα ε, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος προκειμένου να καταλάβουμε είμαι τους δε. Δίχως άλλο, οι καταστάσεις αλλάζουν εύκολα σε ένα κόσμο όπου υπάρχουν πάρα πολλές αναταραχές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε σωστούς στόχους και την κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω ότι η Επιτροπή ε, χρησιμοποίησε μία λέξη κλειδί, ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να έχουν στη βάση τους μία πολιτική. Μία άλλη λέξη που με ευχαρίστησε ιδιαίτερα ήταν η απλοποίηση, η συνοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα. Τώρα που είπαμε ότι ο διάφορος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και συμφωνώ απόλυτα με τους ε, συναδέλφους, ιδιαίτερα με τον συνάδελφο Σάκερ, είπε ότι δεν χρειαζόμαστε τυπικές συναντήσεις, αλλά διαβουλεύσεις. Ο συνάδελφος Κούκαν ε, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία αξιολόγηση από πλευράς της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας αυτού του μέσου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ενιαίο μέσο, πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε, γιατί δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί εδώ. Ας έχουμε μια χαλαρή και προσεκτική στάση. Ήταν πάρα πολύ σημαντική μια παρατήρηση που έγινε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα χωρίς να ξεχνάμε τον όρο δημοκρατία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνάντηση λέγοντας ότι χρειάζονται περισσότερες διαβουλεύσεις για θέματα ουσίας, όχι επίσημες διακηρύξεις και ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε οι μεν τους δε σε ό,τι αφορά τα προγράμματά μας και, και τον τρόπο τον οποίο τα εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ, έχουμε τέσσερις ακόμα ομιλητές, ο χρόνος πιέζει. Ο κύριος Πανσέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομες ε, παρατηρήσεις. Ενώ όλοι μας συμφωνούμε σε ό,τι αφορά το στόχο της καλύτερης διαχείρισης των χρηματοδοτικών μέσων, δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολλές γραφειοκρατικές ε, αντιστάσεις, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες πίεσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε πού οφείλεται αυτή η ανάγκη για ορθολογικό και και θα πρέπει να γίνει μια αναγωγή στην ιστορική μας εμπειρία η οποία θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια καινούργια επιλογή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις. Μια παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα μέσα θα πρέπει να οδηγήσει σε μικρότερη διακριτική ε, ευχέρεια της διοίκησης γιατί πάρα πολλέ φορές στρέφεται κατά της πολιτικής. Ένα παράδειγμα το, το προενταξιακό εργαλείο ενώπιον των δυσκολιών που προκαλούνται από την ελαστική στάση των κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι από τα χρηματοδοτικά μέσα αυτού του μέσου. Δεύτερη σκέψη ελαστικότητα και απλοποίηση. Ναι, μόνο όμως όταν είναι ξεκάθαρες οι πολιτικές προτεραιότητες. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σάριφ όταν ε, λέει ότι θα πρέπει να αποφευθεί μια σύγκρουση μεταξύ της ποσότητας και των προτεραιοτήτων. Αυτή είναι μια πρόκληση πέρα από τις κυβερνήσεις. Η πρόκληση αυτή αφορά το Κοινοβούλιο δεν μπορεί μια πλευρά να ζητά τον έλεγχο ενώ δεν μπορεί να εντοπίσει τις πολιτικές προτεραιότητες, θεωρώντας ότι τα πάντα έχουν προτεραιότητα και με αυτόν τον τρόπο αφήνοντας τα πράγματα ως έχουν. Ενώ για μας υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε κυρίως για να ε, αντιμετωπίσουμε καινούριε προκλήσει μεταξύ των οποίων και αυτή που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι επιλογέ για τι πολιτικέ προτεραιότητε δεν είναι ποτέ ουδέτερο. Το θέμα είναι ποια είναι η ιδέα μα για την Ευρώπη και τι θέλουμε για το μέλλον τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λόπεθ, Στούριθ White. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για το έργο σας, για την έκθεσή σας και την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μέσα είναι μια βασική δράση για την εξωτερική μας ορατότητα, προβολή και για τους πολίτες. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να κάνω δύο ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν τα βλέπω τόσο αισιόδοξα όσο ο Τούνα Κέλεμ. Πόσο ρεαλιστικά ε, θεωρείτε το ενδεχόμενο ε, ε, συγχώνευση των μέσων, όχι ότι συμφωνώ, και το 15% που κρατάτε στην άκρη για μη προγραμματισμένα και έκτακτα, πώς θα γίνει αυτό και πώς θα λαμβάνετε αυτή η απόφαση. Στα ισπανικά θέλω να πω τώρα στο σοσιαλιστή συνάδελφο ότι στο άρθρο 2 ο κανονισμό για το προενταξιακό μέσο δίνει όντω τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα όπως και έπραξε για να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό, να βοηθηθεί, να ανακουφιστεί. Υπάρχει νομική βάση και έτσι νομίζω σωστά, ορθώ έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Sí, muchas gracias. Ο κύριος ε, Γκερέρο, ευχαριστώ. Με κάποια συστολή συμμετέχω σε αυτή την ακρόαση, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών, αλλά την χάνει να είμαι εισηγητής της ίδιας έκθεσης στην Επιτροπή Ανάπτυξης, στο σκέλος που αφορά τα ειδικά μέσα για την ανάπτυξη. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ε, κάνω μερικές ερωτήσεις Ακούσαμε από τις διάφορες τοποθετήσεις ξεκάθαρα ότι υπάρχουν δύο στοιχεία όπου η πολιτική ανάπτυξης και η πολιτική γενική εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ευαισθησίες, ας πούμε ως προς τις αξίες αλλά και τα συμφέροντα. Ή ποιες είναι οι σχέσεις με τους συνομιλητές, με τους εταίρους εκεί επί τους δικαιούχους της ε, αναπτυξιακής μας βοήθειας. Άρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ας απαντήσει όποιος θέλει και όποιο θεσμικό όργανο και όποιος πρόσωπος κοινωνίας των πολιτών. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την ιδιαιτερότητα στα μέσα τα αναπτυξιακά εντός εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αντιλαμβάνεστε ταυτόχρονα την πολιτική ανάπτυξη. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη για πρώτη φορά εγγραφεί στον προπολογισμό και θα μπορεί να επηρεάσει το γενικό μηχανισμό μέσων του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου του επόμενου. Uh, Κυρία Σχάκε, ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ μερικέ ερωτήσει να κάνω, σύντομη θα είμαι όμω, γιατί πολλά τα είπαν οι συνάδελφοι από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε, και ελπίζω να τα σημειώσατε. Κάτι που με εκπλήσει είναι ότι ακούω το εξή από τη μια και με πολύ πιστικά επιχειρήματα και με βάση εκτιμήσει εξωτερικών αναλυτών ότι τα μέσα είναι κατάλληλα για το σκοπό που έχουν σχεδιαστεί. Από την άλλη ακούω ότι χρειάζεται να συγχωνευτούν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Μεγάλο ερωτηματικό, το θέμα της διαχείρισης. Δεν το συζητήσαμε αρκετά ούτε για το πώς μπορεί ε, κανείς γεωγραφικά και θεμετικά να ε, πλοηγητική, ούτε τι κάνει η ΕΔ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διάφοροι ενεχόμενοι που χαίρομαι που ακούσαμε και από την κοινωνία των πολιτών κάποιες ε, απόψεις. Άλλο ερώτημα. Να δοθεί μεγαλύτερη ευθύνη στις ε, επιτόπου αντιπροσωπείες. Βεβαίως είναι πιο κοντά στην πρώτη γραμμή του πυρός, αλλά από την άλλη είναι πολύ μακριά, όσο γίνεται μακρύτερα από εμά, από την αναθεώρηση, από τον έλεγχο και μπορεί να έχουμε σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων ε, υπάρχει ανάγκη να έχουμε και ρεαλιστική σχέση με την κυβέρνηση μιας χώρας από τη μια και από την άλλη να ε, βοηθήσουμε τις πιο σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό πώς θα το κάνουμε και πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο χωρίς να έχουμε τριβές και συγκρούσεις. Έχω και μια ερώτηση του David McAllister να επαναλάβω πριν φύγει. Για ποιο λόγο δεν έχετε καταθέσει κάτι εξοδότηση πράξης. Δεν έχετε απαντήσει σε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνοψίζω λοιπόν. Πολύ ε, αναφέρατε ότι ορισμένες από τις βασικές αρχές ε, είναι πιο ευπρόσδεκτες, να είμαστε πιο προσανατολισμένοι στην πολιτική και όχι στο μέσο, να είμαστε πιο ευέλικτοι. Αναφερθήκατε και σε συγκεκριμένε ε, ανησυχίες, ότι ο διάβολος κρύβεται στι λεπτομέρειες, ότι χρειάζεται έλεγχος, εποπτεία, χωρίς συμβιβασμού και χωρίς να διακυβεύονται όλα αυτά. Λεπτομέρειες δεν άκουσα όμως για τη διακυβέρνηση ιδιαίτερα και πώς όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Μπορεί να μην ε, είστε σε θέση να απαντήσετε σε όλα αυτά σήμερα, αλλά οι απαντήσει αυτές χρειάζονται πριν προχωρήσουμε συγκεκριμένα και από ό,τι ακούτε υπάρχουν πολλές ανησυχίες από πολλές πολιτικές ομάδες. Έχουμε ένα δεκάλεπτο χονδρικά. Άκουσα ότι μας δώσανε και άλλο χρόνο. Προσωπικά πρέπει να φύγω όμως. Οπότε θα χρειαστεί ίσως να προεδρεύσει κάποιος άλλος. Α, χαίρομαι που έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Ποιος θέλει το λόγο, Κρίστιαν. Um, Με χαρά να ξεκινήσω, ο κύριος Λεφλέρ. Και σας ευχαριστώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θέλω να προκαλέσω τώρα μερικού από του ομιλητέ και από του βουλευτέ. Με εκπλήσει ο συντηρητισμό σα. Μιλήσαμε για το διάβολο και τις λεπτομέρειες. Αλλά βλέπω και κάποια επανάπαυση στη βολή μας. Δηλαδή, καλός είναι ο διάβολος που γνωρίζουμε και όχι το καινούριο. Για τις κατεξοδότηση πράξεις. στην όλη αρχιτεκτονική όταν σχεδιάστηκε η οποία αποφασίστηκε σε συναπόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το σημερινό PDP, το κάθε μέσο χωριστά τεχνικά είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Λειτουργούν αυτά. Ε, διαχειριζόμαστε ε, τις καταστάσεις που πρέπει. Κάνουμε τη δουλειά για την οποία έχουν σχεδιαστεί. Και μετά καταλήξαμε με τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει λόγος να ανασχεδιαστεί όλο αυτό το οικοδόμημα εκβάθρων. Και στην ενδιάμεση αναθεώρηση δεν διαπιστώσαμε την ανάγκη να μετατοπιστεί ε, καμιά τεράστια πρικοδότηση από μια χώρα ή μια περιφέρεια σε μια άλλη. Γιατί και αυτό θα χρειαζόταν κάτι εξουδότηση πράξη. Τη στιγμή που σχεδιάστηκαν λοιπόν τα μέσα υπήρξε ένα περιθώριο για τέτοιου είδους μετατοπίσεις για ποσά σε επίπεδο που θεωρήσαμε εμείς υπαρκές. Κατά τα άλλα αντιλαμβάνομαι ότι τα έγγραφα για τη συζήτηση για τη στρατηγική αναθεώρηση έχουν διαβιβαστεί σήμερα που θα γίνει εδώ αυτή η συζήτηση. Έχετε τρεις εβδομάδες για να τα κοιτάξετε, για να κάνετε και ερωτήσεις, για διευκρινήσεις κτλ. Για ποιο λόγο λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι εφόσον λειτουργούν καλά για περισσότερη ε, εδραίωση και ενίσχυση. Γιατί μπορεί, χωράει βελτίωση αρχιτεκτονική για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και το πιστεύουμε. Και μάλιστα απλουστεύοντας τις διαδικασίες θα μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε περισσότερο και να εστιάσουμε στα σημαντικά, στην εκάστοτε πολιτική και τους στόχους της. Εκεί θα πρέπει να αφιερώσουμε την προσοχή μας. Όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά ε, με μια συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την επόμενη γενεά μέσων, ήταν παλιά βέβαια, δεν πολύ θυμάμαι, αλλά είχαμε πάνω από 20 μέσα για τις εξωτερικές σχέσεις. Μέχρι σήμερα αυτά έχουν γίνει τα μισά, έχουν μείνει 10. Πάνω κάτω εσωτερικά, εξωτερικά δεν θεωρούμε ότι σήμερα είναι λιγότερος ο έλεγχος από εκείνο που υπήρχε πριν από 15-20 χρόνια. Πιστεύουμε ότι έχουμε αυξήσει την αποτελεσματικότητα και έχουμε προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Η εδραίωση, ε, η ισχυροποίηση έχει να κάνει με τη διαχείριση, με τις δομές και τις λειτουργίες. Δεν πρόκειται να προτείνουμε ένα μοναδικό στόχο πολιτικής. Βεβαίως, τέτοιο ερώτημα τι θα γίνει αν εγγραφεί στον προπολογισμό το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, τι θα γίνει με την αναπτυξιακή πολιτική. Μα το είπαμε πέρσι, ανανεώθηκε η συνένεση που επιτρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών και με ε, την ατζέντα του 2020 να το εντάξουμε. Αυτό είναι το πολιτικό μας πλαίσιο. Από εκεί και πέρα πώς θα γίνουν αυτά διαδικαστικά. Είναι τεχνικά ζητήματα περισσότερο. Και προφανώς θα βγουν διάφοροι διαβολάκια στις λεπτομέρειε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε με μια πιο απλοποιημένη δομή διατήρησης να διατηρήσουμε διαχείριση συγγνώμη, και τη θεματική μας ε, διάσταση και τη γεωγραφική διάσταση και τη διάσταση της άμεσης δράσης που είναι σημαντικά αυτά χωρίς να αποδυναμωθεί τίποτα με κοινή κινητοποίηση για τον ίδιο στόχο. Εξού και η ευελιξία. Και κάποια άλλη ευελιξία που ακούστηκε επανελειμμένα είναι τι κάνουμε με τις επιδόσεις. Ο κύριος Κούκαν ρώτησε. Αναφέρθηκε στην αρχή more for more, Περισσότερο για περισσότερο. Αυτό ήδη ισχύει σε αρκετά μετροπαθές επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό. Το να δίνεις περισσότερα χρήματα ανάλογα με τις επιδόσεις, δεν αλλάζει και τίποτα γιατί είναι μικρό το ποσό. Άρα στο μέλλον θα πρέπει να εμπνευστούμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για να βελτιώσουμε την αρχιτεκτονική όπου υπάρχει ένα αποθεματικό και μεγάλο για έκτακτα, απρόοπτα γεγονότα, μη προγραμματιζόμενες δαπάνες που είναι πολύ συχνό αυτό ακριβώς για να μπορέσουμε να υποστηρίζουμε εκείνους από τους εταίρους μας που πραγματικά καταβάλουν προσπάθεια. Και αν κάνουν εκείνη τη διαφορά θα ανταποκριθούμε κι εμείς. Αυτό είναι το σκεπτικό και η λογική που λέει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα σεβαστό ποσό, σε αποθεματικό στην αρχή, χωρίς να έχει εγγραφεί προγραμματισμένο με στρατηγικό διάλογο και με προοπτική για το μέλλον να δούμε ποιες είναι οι ε, προτεραιότητες σε ένα τοπίο μεταβαλλόμενο. Τι ρόλο έχουν να παίξουν τώρα οι αντιπροσωπείες μας επί τόπου και πώς μπορούμε να αναθέσουμε σε εκείνες τη διαχείριση. Νομίζω το ερώτημα αυτό είναι ψεύτο ερώτημα γιατί τελικά η διαχείριση της βοήθειας μας εντάσσεται γράφεται σε ένα τρίγωνο που θα πρέπει να λειτουργεί κάθε πλευρά, η κάθε γωνιά του τριγώνου. Δηλαδή η διαχείριση με την καθοδήγηση του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Είναι τρίγωνο. Και εσείς είστε πάνω από το τρίγωνο. Ε, τρει, τρεις πλευρές του τριγώνου ή τρεις γωνίες είναι η Γενική Διεύθυνση Αρμόδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι διαχειριστικές αρχές, κατά τόπους υπηρεσίες και η τρίτη γωνία είναι οι αντιπροσωπείες τόπου. Άρα, θα πρέπει να δούμε πώς οι στρατηγικές κατευθύνες γραμμές που λαμβάνουμε από εσά και από τα κράτη-μέλη θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους για να δούμε πώς το πρόγραμμα αυτό θα γίνει συγκεκριμένο έργο. Project. Αλλά οι προσωπίες μας εκεί στις διάφορες χώρες θα μας βοηθήσουν να τα μεταφράσουμε αυτά στην πράξη. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε ωραίες ιδέες και σχέδια, αλλά πώς αυτά στην πράξη μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό θα αποφασίσουν εκείνοι, θα μας βοηθήσουν και θα έχουν τη δική μας στήριξη. Και όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, χρειάζονται την στηρίξει για να έχουν και το θάρρο να αντιμετωπίσουν δύσκολε καταστάσει. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία των πολιτών, όπου χρειάστηκε ή χρειάζεται να κάνουμε μια εξαίρεση σε αυτό το μοντέλο του τριγώνου γιατί κάποια από τι γωνίες σε περίπτωση αυτή θα ήταν υπερβολικά εκτεθειμένοι. ή οι εταίροι μας, οι δικαιούχοι. Πάντως αυτή η τριγωνική σχέση θα πρέπει να είναι αποτελεσματική κάθε ε, πλευρά του τριγώνου να κάνει τη δική του της δουλειά και μετά θα ερχόμαστε σε εσά. Ελπίζω να έχουμε επιτύχει να μεταφράσουμε τις δικές σας προτεραιότητες σε συγκεκριμένη δράση. Ευχαριστώ Κρίστιαν. Νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει μια μακρά συζήτηση και για την ομάδα εργασίας των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων θα κάνουμε μια συνάντηση στα θέματα της διαχείρισης και στις ανησυχίες οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια για την ανάγκη που υπάρχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καθοδηγεί τη διαδικασία έτσι ώστε να αποφύγουμε μια σκοτεινή δομή όπου κανένας δεν θα γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνο και γιατί. Για την έκθεσή μου η 7η Φεβρουαρίου 11η πρωινή είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ανταλλαγή απόψεων στις 21 ή 22 Φεβρουαρίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 20 Μαρτίου. Έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, όπως επίσης και τα Think Tank, τους αξιολογητές και εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας και τον χρόνο σας. Αφήτα.